πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας κατάσταση στην Ιεμένη. Ο Επίτροπος Χάν έχει εκ νέου το λόγο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσω μαζί σας εξ ονόματος της Φεντερίκα Μογκερίνη όσον αφορά την κατάσταση στην Ιεμένη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ σημαντική κρίση στη Μέση στην Ανατολή, αλλά στα πλαίσια της κρίσης αυτής θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την κρίση στην Ιεμένη. Η Ιεμένη, η Ιεμένη κατέχει μια στρατηγική θέση στον κόλπο του Άντεν και βρίσκεται πολύ κοντά στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και πραγματικά βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί προς την Ινδικό ωκεανό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κρίση στην Ιεμένη ενδεχομένως να επηράσει την ε, ευρύτερη γύρω περιοχή. Επίσης, ε, οι εξελίξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη καταδεικνύουν ότι αυτή τη στιγμή τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η ISIS και η Al-Qaeda στην Αραβική Χερσόνησο εκμεταλλεύονται το κενό εξουσίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη προκειμένου να ανακτήσουν έδαφος και ισχύ. Και αυτό αποτελεί απειλή και κίνδυνο για όλες τις χώρες περιοχής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό στα πλαίσια της κοινή εξωτερικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά θα πακολουθήσει χάος. Μετά την 4η Ιουλίου συμπληρώθηκαν 100 μέρες από τότε που ο επικεφαλής της χώρας Χάντι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα της χώρας της Σανά και από τότε που είδαμε ότι οι ΣΥΙΤΕΣ αντάρτες Χούτι άρχισαν να προλάβουν προς το, προς το νότιο της χώρας. 14.000 είναι 3.000 συνεκροί και ένα 80% του συνολικού πληθυσμού βρίσκεται σε πήγους ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας εν μέσω επισητιστικής κρίσης η οποία εκτελήσεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα άτομα που χρειάζονται βοήθεια στην Ιεμένη ε, από ότι στο σύνολο της περιοχής νοτίως του Σαχέλ. Πρέπει λοιπόν, όπως ακριβώς φαίνεται και στα συμπεράσματα του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου του ε, 2015 να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες δράσεις. Έχουμε επίσης συγκεκριμένη δήλωση της ΥΠΑ εκπροσώπου και του Επιτρόπου Στυλιανίδη όσον αφορά την επίλυση της υφιστάμενης κρίσης, η οποία επίλυση μπορεί να περάσει μόνο μέσω από συζητήσεις που θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια των ΗΕ και μέσω επικοδομητικού διαλόγου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Υπάρχουν συγκεκριμένα ψηφίσματα των εθνών τα οποία δεν έχουν γίνει σεβαστά και αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Ξέρετε ότι τα ψηφίσματα των εθνών έχουν θέσει συγκεκριμένε παραμέτρου και συγκεκριμένα το ψήφισμα 32 32-6 θα μπορούσε να επιφέρει μια λύση για την κρίση, αντιμετώπιση των τρομοκρατικών οργανώσεων και παρεμπόδιση οποιασδήποτε περαιτέρω περιφερειακής αστάθειας. Ξέρετε ότι ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, υπάρχει μια κρίση που έχει μια έντονη πτυχή κοινωνική, οικονομική, πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή τη στιγμή όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Από τις 15 στις 20 Ιουνίου έγιναν συζητήσεις στην ε, Γενέβη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πολιτική αποκατάσταση στη χώρα. Έχουμε μια πολύ θετική προσέγγιση από τον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έθεσε τις βασικές προϋποθέσεις για να πάυσουν οι διαμάχες και να οδηγηθούμε σε μια εκεχηρία. Και θα πρέπει βέβαια να ε, προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στις βασικές κεντρικές πόλεις της Ιεμένης. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε όλους τους διαπλεκόμενους, όλες τις αντιμεχόμενες πλευρές και θα πρέπει βέβαια να συμβάλλουν ακόμα και οι σύντες αντάρτες Χούτι. Θα πρέπει να ακολουθηθούν όμως οι παράμετροι που έχουμε στο ψήφισμα των ΗΕ Εθνών υπαριθμών 2260. Θα πρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη λοιπόν να συμβάλλουν στη διαδικασία που προβλέπεται από την ΗΕ καλή την πίστη. Και κατά αυτόν τον τρόπο όλες οι ανησυχίες που έχουν προκύψει θα ληφθούν υπόψη στα πλαίσια μιας ευρύτερης πολιτικής ε, λύσης και διευθέτησης. Η ανθρωπιστική κρίση από τις ε, συνεχόμενες αυτές διαμάχες και από, τις, ε, από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς πλήττει ιδιαίτερα τους πολίτες και ιδίως τα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει πραγματικά σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα όσον αφορά στην κρίση αυτή. Μιλάμε για μια πραγματική σοβαρή, σοβαρότατη ανθρωπιστική κρίση. Οι υποδομές της χώρας βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό συμβαίνει ακόμα και για τις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Σε ένα τέτοιο λοιπόν μετάβλητο περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει πραγματικά στους πολίτες Ιεμένης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθαν υποστήριζε τις προσπάθειες των Εθνών για να έχουμε μια βιώσιμη, προβλέψιμη ε, η οποία θα σέβεται την ανθρωπιστική διάσταση και θα επιλύει την ανθρωπιστική κρίση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την παροχή τροφίμων, καυσίμων καθώς επίσης και κάποιων βασικών αγαθών και προϊόντων η οποία θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ουδέτερο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρόσβαση στην Ιεμένη για το εμπορικό ναυτικό να διευκολυνθεί και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των ΕΕ 2260 κατά τρόπο αναλογικό και προβλέψιμο. Επίσης θα πρέπει να γίνουν και επιθεωρήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει επιτόπου να επιβλέψουν όλες τις διαδικασίες, ιδίως εκείνες που αφορούν την παροχή τροφίμων και καυσίμων με πλοία δια της θαλάσσης μέσω της Ιεμένης. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να γίνει σεβαστό το ανθρωπιστικό δίκαιο και να προστατεύσουμε τους πολίτες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση καμία από τις δύο πλευρές να βάλει κατά των ίδιων των πολιτών ή κατά των υποδομών εκείνων που εξυπηρετούν τους πολίτες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σημαντικές υποδομές όπως νοσοκομεία για, από το στρατό ή για στρατιωτικούς λόγους. Χρειαζόμαστε επίσης ομάδες διάσωσης, χρειαζόμαστε νοσηλευτικό προσωπικό και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μπορούν να φτάσουν ασθενοφόρα καθώς επίσης και φορεί παροχή υγειονομικών υπηρεσιών στι πιο ευαίσθητε περιοχέ. Το Ανθρωπιστικό Γραφείο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ΕΚΟ, έχει ήδη κινητοποιήσει 25 εκατομμύρια ευρώ για την Ιεμένη, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι επίγουσε ανάγκε τη χώρα. Διπλωματικέ όμω προσπάθειε γίνονται επίση, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση όλων των, όλου του ανθρωπιστικού προσωπικού προς όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια να συνειδητοποιήσουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα ευοδοθεί αν δεν καταφέρουν τα πλοία διαθαλάσσης να φτάσουν στην Ενιεμένη και να φέρουν αυτό το 80% των συνολικών προϊόντων που προβλέπω ότι θα πρέπει να δοθούν ως ανθρωπιστική βοήθεια στην Ιεμένη. Η λύση στην κρίση αυτή θα πρέπει να είναι σαφώς πολιτική και κάθε μέρα που περνάει μας ε, βυθίζει όλο και περισσότερο στην πόλωση και πολύ φοβόμαστε ότι κάθε μέρα που περνάει χωρίς δράση μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ πιο έντονη διένεξη και αντιπαράθεση. Υποστηρίζουμε λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα Ηνωμένα Έθνη και θέλουμε να πείσουμε όλες τις πλευρές να κινηθούν γρήγορα στο δρόμο της ειρήνης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή για να ακούσω τις απόψεις σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ας ξεκινήσει λοιπόν τώρα η συζήτηση. Δεν είμαστε πάρα πολύ στην αίθουσα αυτή, αλλά η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να καλωσορίσω και κάποιους επισκέπτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το λόγο έχει πρώτα η κυρία Λιώ Μαρή για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το η Γεμένη σήμερα αποκρισταλώνει τις περισσότερες εντάσεις και αντιπαλότητες που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Ο περσικός κόλπος θα μπορούσε να χάσει την ισορροπία την γεωστρατηγική όπως τονίσατε και οι ανισορροπίες στον κόλπο θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις πάνω στο σύνολο της Μέσης Ανατολής και στις χώρες δίπλα στον κόλπο του Άντεν. Και ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτή η αποσταθεροποίηση δεν θα είχε αντίκτυπο στη δική μας κατάσταση, είτε πρόκειται για την οικονομική κατάσταση ασφαλείας ή πολιτισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί λοιπόν να αδιαφορήσει για αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα που είναι απομακρυσμένη, που δεν είναι καλά γνωστή όπως το διαπίστωσα, διότι αυτή μπορεί να έχει επιπτώσεις στις χώρες μας. Σήμερα η Σαουδική Αραβία και οκτώ αραβικές χώρες, Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Ιορδανία, Κοβέιτ, Μαρόκο, Κατάρ, Σουδάν και τα Εμμυράτα με την υποστήριξη της δυτικής κοινότητας έχουν μια κοινή επιχείρηση στρατιωτική ε, για να αντιτεθούν στους Χούτι και στον Τάσ. Οι χώρες αυτές που έχουν ε, εχθρό τις αντιπελότητες μεταξύ τους έχουν συνασπιστεί για την ίδια επιχείρηση. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ισορροπία, την ισορροπία που χρειάζεται για την περιφερειακή σταθερότητα. Μην ξεχνούμε ότι οι χώρες του κόλπου είναι οι πρώτοι συμμαχοί μας στον καταπολέμηση του Νταέσ και της ε, τρομοκρατίας. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια για να συμμετάσχει στην αποκατάσταση σταθερότητα στην Γεμένη. Δεν αρκεί να υποστηρίξουμε τη μία ή άλλη πρωτοβουλία διότι εμείς ε, δεν έχουμε ε, χρηματοπιστωτικά και οικονομικά συμφέροντα στη χώρα, μπορούμε ε, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Τι κάνουμε για να υποστηρέξουμε τους άμαχους ε, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που πλήττονται και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πρόκειται να λάβετε πρωτοβουλίες για να δημιουργήσετε μια νέα κατάσταση για τις γυναίκες στη χώρα αυτή, για τις οποίες γίνεται λίγος λόγος, αλλά οι οποίες έχουν το καθεστώς ε, το πιο λυπηρό του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χάουιτ έχει τώρα το λόγο εξ ονόματων των Σαλιστών για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σε αυτή τη συζήτηση κυρίως ασχολούμεθα με την μεγάλη καταστροφή, ανθρωπιστική καταστροφή που λαμβάνει η χώρα στην Ιεμένη. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν διακηρύξει μια ανώτατου επίπεδου τέτοια, ε, ένα τέτοιο συναγερμό για την ανθρωπιστική αυτή καταστροφή ο πληθυσμός 1,5 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από ασυτεία και ακόμα περισσότερα εκατομμύρια έχουν προσθεθεί σε αυτήν την κατάσταση πρόσφατα. Βρίσκεται η Ιωεμένη μία, ένα βήμα από τη λιμοκτονία. Ένα, ε, τα ποσά που δόθηκαν δεν ήταν αποτελεσματικά και βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι τα κυριότερα θύματα. Το ψήφισμά μας τίθεται υπέρ της ανθρωπιστικής αυτής υποστήριξης, υποστηρίζοντας ε, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η ομάδα μου <clears throat> τοποθετείται ενάντια σε όλες αυτές ε, τις ε, επιθετικές πράξεις ε, και όσον αφορά τις, τους Χούτις και τις, των Αλφαγιές και οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις των βομβαρδισμών και του αποκλεισμού από τη Σαουδική Αραβία και τη Συμμαχία είναι κάτι που καταγγέλουμε. Η νομιμότητα της στρατιωτικής παρέμβασης από πλευράς του πρώην Προέδρου όταν είχε ήδη παρετηθεί <clears throat> δεν καθιστά καθόλου περισσότερο νόμιμη την κατάσταση αυτή σε σχέση για παράδειγμα με τον Ουκρανό πρόεδρο Γιαννουκόβιτσα αλλά σε ένα άλλο πλαίσιο αυτό. Και η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών με το άρθρο 51 που αφορά την ε, ε, προστασία της χώρας από εξωτερικούς εχθρούς δεν μπορεί να νομιμοποιήσει αυτές τις πράξεις και βλέπουμε ότι ε, πρέπει όλοι να συμμετάσχουν για την σταθεροποίηση της περιοχής. Ζητούμε να πάψουν οι διώξεις όσον αφορά τις θρησκευτικέ πεπιθήσεις και Επίσης πρέπει να πούμε ότι πρέπει να δούμε τον ε, μεγάλο ρόλο που διαδραματίζουν εδώ οι ακραίοι Ισλαμιστές όσον αφορά την πιο φτωχή αυτή χώρα. Είναι λοιπόν ε, άμεσα, άμεση η στόχη αυτού του ψηφίσματος να σταματήσει η βία Όλες οι προσπάθειες πρέπει να στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση για μια υποδιαπραγμάτευση ειρήνη, ώστε να πάψει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματος του ECR, ο κύριος Τάνοκ τώρα για ένα λεπτό. Κύριε... Πρόεδρε, η, Εμένη δείχνει τι επήγε στραβά σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη, με τον τότε πρόεδρο Σαλέχα και την χώρα εκείνη που πραγματικά έχει υποστηρίξει τους Χούτης και τη Σαουδική Αραβία που υποστηρίζει τους αντιπάλους που βρίσκονται τώρα στο Ριάντ. Χρησιμοποιείται η στρατιωτική βία όσον αφορά τους ε, προηγούμενους οπαδούς ε, του Προέδρου Σάλε. Η χώρα αυτή έχει γίνει μια ζώνη ανθρωπιστικού ολέθρου πάνω από το ίμιση των αμάχων, γυναίκες και παιδιά υφίστανται τα πάνδυνα από, τις, ε, από τους βομβαρδισμούς ε, όσον αφορά την εκλεγήσα κυβέρνηση Χάντι. Υπάρχουν καταγγελίες ε, για παραβιάσεις, κατάφορες παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και βλέπουμε το τι συμβαίνει στον κόλπο του Άντεν και τις δράσεις της Αλκάιντα στην Χερσόνησο της Αραβίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μεγάλο ρόλο πέρα από την υποστήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας και φυσικά καλώ όλες τις πλευρές να επανέλθουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και να πάψουν οι εχθροπραξίες. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε. Κύριε Τάνοκ. Ε, υπάρχει μια ερώτηση για σας εξ ονόματος του κυρίου Κάρμπερ. Τη δέχεστε? Πολύ ωραία. Κύριε Κάρμπερ, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Τάνοκ που δεχτήκατε την μπλε κάρτα. Υπάρχουν προφανώς πολιτικές διαφορές, αλλά συμφωνείτε με αυτό το οποίο θα πω, να υποστηρίξουμε την Σομαλιλάνδη και να αναγνωρίσουμε τη Σομαλιλάνδη που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του κόλπου του Άντεν και να βοηθήσουμε βασικά και τους πρόσφυγες οι οποίοι προέρχονται, που έχουν πάει Σομαλιλάνδη από την Ιεμένη. Ναι, όντως πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναγνωρίσουμε τη Σομαλιλάνδη. Είναι δημοκρατική, έχει το κράτος δικαίου ως βασική αρχή και έχει συμβάλει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της πειρατείας και του Ισλαμικού, της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Ήταν Βρετανικό προτεκτοράτο στο παρελθόν, ονομαζόταν τότε Βρετανική Σομαλιλάνδη και Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε αυτό το οποίο είπατε. Βέβαια, η σημερινή συζήτηση δεν έχει να κάνει με τη Σομαλιλάνδη αυτή καθεαυτήν, μόλον το ζήτημα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η σημερινή συζήτηση έχει να κάνει με την κατάσταση στην Ιεμένη. Και προφανώ υφίσταται μια ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή, όπω είπα και στην παρέμβασή μου, και υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγε που όντω διέσχισαν το κόλπο του Άντεν και έχουν πάει στην Σομαλιλάνδη στην Βαρβέρα συγκεκριμένα, στο λιμάνι της Βαρβέρας. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να γνωρίσουμε τις προσπάθειες της Σομαλιλάνδης, η οποία έχει υποδεχθεί πάρα πολλούς τέτοιους πρόσφυγες. Ευχαριστούμε πολύ. κυρία Σάκια έχει τώρα το λόγο για δυόμιση λεπτά. Παρακαλώ. Εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Οι φτωχοί πολίτες της Ιεμένης πάσχουν από την απουσία ενός μιας δημοκρατικής κυβέρνησης και από την ένταση και τις βιοπραγίες κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Χιλιάδες έχουν δολοφονηθεί και ακόμα πολύ περισσότεροι τραυματίστηκαν στις τελευταίες εκρήξεις βίας που ξεκίνησαν την άνοιξη του 2015. Υπάρχουν εκθέσεις ότι η συμμαχία υπό την Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς και θα πρέπει να εξεταστεί αυτή η καταγγελία από τα Ηνωμένα Έθνη και πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες κυρώσεις και επιπτώσεις αληθεύει αυτό. Και οι διακριβώσεις και ανακρίσεις πρέπει να εξετάσουν και άλλα εγκλήματα που έχουν καταγγελθεί για να δούμε κατά πόσον αυτά είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και βλέπουμε ότι χρειάζεται η αποκλιμάκωση της βίας για να επανασταθεροποιηθεί η χώρα. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή και τα δεινά τα οποία υφίστανται οι πολίτες πρέπει να σταματήσουν. Ζητούμε από όλους που εμπλέκονται σε αυτές τις σειράξεις να σταματήσουν τη χρήση της βίας. Ενώ οι πολίτες υφίστανται τα πάνδυνα, η Αλκάιντα, το Ισλαμικό κράτος και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις ε, εποφελούνται και αυξάνονται μέσα στο χάος της Ιεμένης οι προσπάθειες για την ανθρωπιστική βοήθεια μέσα από αυτές τις βιοπραγίες πραγματικά στραγγαλίζονται και βλέπουμε μια τοξική σπυροειδή εξέλιξη προς τα χειρότερα και στρατολογούν παιδιά για τις δραστηριότητες τους οι τρομοκράτες ε, και αυτό είναι κάτι που πραγματικά μας κάνει να ντρεπόμαστε. Πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν με κάθε τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ο διάλογος και η αποκλιμάκωση της βίας και να αναζητηθεί μια πολιτική λύση στα πράγματα συμπεριλαμβανομένου και ενός πιο επικοδομητικού ρόλου των ε, περιφερειακών εταίρων που όπως επεσήμαναν οι συνάδελφοι εμπλέκονται ιδιαίτερα στην κατάσταση της Ιεμένης και αυτό οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη βία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τις εταιρικές σχέσεις που έχει και συμφωνίες με κάποιες χώρες εταίρους σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής οι αλλοδαποί ε, ε, εμπλεκόμενοι πρέπει να σταματήσουν αυτές τις εχθροπραξίες. Και εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξουμε οποιασδήποτε προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για έναν πολιτικό διάλογο και ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω και να είναι προπομπός, πρωτοπόρος σε αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ο κύριος Κούζο Περμού για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια σύραξη, σε μια σύγκρουση που προκαλεί τεράστια δεινά και είναι υποδειγματική η κατάσταση αυτή για τη δημιουργία χάους στη ζώνη αυτή. Το χάος αυτό που έφτασε ε, με τους πολέμους ε, ε, μέσω εντολής άλλων εμπλεκόμενων. Και πραγματικά παρατηρούμε απλά και μόνο πως ε, μια συμμαχία από την, υπό την Σαουδική Αραβία, μια δικτατορία θεοκρατική που είναι και σύμμαχός μας, ε, που βομβαρδίζει με απαγορευμένα όπλα τους αμάχους και έχει αποκλείσει με ναυτικό αποκλεισμό, πράγμα το οποίο υφίστανται τα πάνδυνα οι πολίτες, οι άμαχοι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει στρατιωτική λύση λοιπόν. Γι' αυτό ζητούμε μια ολοκληρωμένη πολιτική λύση, την κατάργηση του ναυτικού αποκλεισμού το σταμάτημα, την πάυση των βομβαρδισμών και να μπορέσει η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία να επιμείνουν όσον αφορά τον κώδικα εξαγωγής όπλων να τηρούνται διαδικασίες. Ευχαριστώ. Σμιτ παρακαλώ. Κύριε Πίτροπε, ε, σημερίζουμε τα σχόλιά σας ότι η μακροπρόθεσμη λύση θα μπορούσε να λύσει την κατάσταση. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη σύγκρουση στην Γεμένη, διότι αυτό βοηθάει μόνο τους εξτρεμιστές και δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος γι' αυτό, Σχετικά με το τι πρέπει να γίνει βραχυπρόθεσμα, ούτως ώστε οι προσπάθειες οι ανθρωπιστικές να μπορούν να αποδώσουν, Υποστηρίζω ότι χρειάζεται μια διακοπή ούτως ώστε να προωθηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά πρέπει να δούμε, να ελέγξουμε τον συνασπισμό των Σαουδαράβων. Πάρα πολλές ε, κυβερνήσεις βοηθούν ε, την, ε, αυτήν την παρέμβαση και η τακτική είναι αμφισβητήσιμη η νομιμότητα της ε, επιχείρησης αυτής ε, συζητείται και θα πρέπει να ελέγξουμε την επιχείρηση αυτή διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίζεται και να υποφέρει ο λαός της Γεμένης και εμείς ε, απλώς να παρακολουθούμε. Εξ ονόματος του FDD ο κύριος Κάρπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες είχαμε μια ομάδα, ε, τα διάφορες πολιτικές ε, ομάδες που θέλουν ε, να επανέλθουν στα σύνορα πριν από το 1990. Ο ε, αντιπρόεδρος της Νοτίου Γεμένης μας έδωσε μια εικόνα, μίλησε με πάθος για την, ε, για την αύξηση της ανθρωπιστικής κρίσης, το, το ότι η βοήθεια ε, διανέμεται με περίεργο τρόπο δεν αποφέρει το, το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι είναι αναλφάβητοι, είναι θέματα πιεστικά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, να υπάρξει εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός, ούτω ώστε να μπορούμε να ασχοληθούμε με το ανθρωπιστικό θέμα ως θέμα προτεραιότητας. Θα πρέπει κατεπηγόντως να ασχοληθούμε με το θέμα να, και ίσως δεν αντιπροσωπεύουμε τις οργανώσεις που και τα κινήματα της νότιας κίνησης είναι στο τραπέζι και ζητούν, μα ζητούν να δράσουμε για αυτούς. Ο κόσμος λοιπόν ε, ε, έχει δέχεται αυτό τον διχασμό ανάμεσα στους Σουνίτες και στους Σίτες. Η Γεμένη είναι παράδειγμα αυτού του διχασμού. Δεν θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να θεωρήσει αν ε, η ενωμένη Γεμένη είναι κάτι το βιώσιμο. Ίσως τελικά θα πρέπει να διαιρεθεί η Γεμένη ε, στα σύνορα πρώτης ενοποίησης. Δεν έχουμε μάθει τίποτα από τα σφάλματα που έγιναν πριν από έναν αιώνα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τις ομιλίες από τις πολιτικές ομάδες. Περνάμε στους μονομένους τώρα ομιλητές με πρώτον τον κύριο Ποσπισίλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Τη συζήτηση αυτή την παρακολούθησα εκ του σύνεγγυς πολύ προσεκτικά. Άκουσα τι είπε ο Επίτροπος και ευχαριστώ για αυτό, για το ότι εδώ σήμερα απόψε στην Ολομέλεια ασχολούμεθα με αυτό το θέμα. Έχουμε αυτή τη συζήτηση για την κατάσταση στη Συρία, στο Ιράκ, εξάλλου και πολύ συχνά η κατάσταση όσον αφορά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ιεμένη ξεχνάμε το τι συμβαίνει εκεί. Όμως πρόκειται για μια περιοχή που έχει στρατηγικά τεράστια σημασία και εφόσον αυτός ο εμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αντιπαράθεση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών. Και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα επικίνδυνο. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ώστε να οδηγήσουμε σε μια αποκλιμάκωση αυτής της βίας. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε την κατάσταση ήδη σύντομα και όλας να την αντιμετωπίσουμε θετικά. Έχω κάποιες επιφυλάξεις, αλλά τουλάχιστον να αναχαιτήσουμε τη βία. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, να την μειώσουμε. Και εξάλλου οι τρομοκρατικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ιεμένη ενισχύονται περαιτέρω με αυτή την κατάσταση. Μια αποδυνάμωση της κεντρικής κυβέρνησης στην Ιεμένη ταυτόχρονα ενδυναμώνει από την άλλη πλευρά την Αλκάιντα και το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Συρίας. Είναι ένα σενάριο το οποίο μας κάνει να φοβόμαστε ιδιαίτερα. Γι' αυτό ζητούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδυναμώσει τον πολιτικό διάλογο. Ιδιαίτερα όμως να προσπαθήσει την ανθρωπιστική κρίση σε αυτή τη χώρα που αφορά μυριάδες να την αντιμετωπίσει. Όλα. Για ένα λεπτό κύριο κύριος Καν. Κύριε Πρόεδρε, μετά από 100 μέρες ε, όσον αφορά τη διένεξη αυτή βλέπουμε ότι η κατάσταση ανθρωπιστική επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Έχουν χαθεί πάρα πολλές ζωές στη διένεξη αυτή. Και ανησυχώ τώρα πάρα πολύ ότι ε, ενώ η βία μπορεί τελικά να γίνει περιφερειακή διένεξη, αυτή με τη σειρά τη θα αποσταθεροποιήσει περισσότερο τη Μέση Ανατολή και θα πλήξει όμω ακόμα και τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ηθική υποχρέωση να βοηθήσει την Ιεμένη και το λαό τη. Πρέπει λοιπόν καταρχά να σταματήσουμε τη βία. Θα πρέπει να έχουμε μια ανθρωπιστική εκεχηρία προκειμένου να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στο 80% του πληθυσμού τη χώρα. Αλλά μπορεί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν συνεργαστεί η Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Η βασική περιφερειακοί παράγοντες πρέπει να αναλάβουν ευθύνη προκειμένου να βοηθηθεί ο λαός της Ιεμένης. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, την ανεργία, την απουσία των βασικών υπηρεσιών που πραγματικά έχουν συμβάλει στην ανθρωπιστική κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη. Εμείς θεωρούμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταθλητές όσον αφορά τις ε, κοινωνικές, οικονομικές υπηρεσίες. Οφείλουμε λοιπόν να τις προσφέρουμε για να βοηθήσουμε το σύνολο των πολιτών της Ιεμένης. Σας ευχαριστούμε πολύ για ένα λεπτό κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε ο χάος και η σύγκρουση στην Ιεμένη είναι σαν μια ε, σπυροειδής ε, κλιμάκωση και καλύπτονται και οι Λιβύοι και άλλες χώρες ε, οι οποίες ολίστησαν σε αυτού του είδους τη σύγκριση. Είναι χώρες που έχουν αποτύχει. Ο συνασπισμός και η επιχείρηση δεν επιτυγχάνουν τίποτα. Επίσης παρακολουθούμε μια επιβράδυνση στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων με επικεφαλής τον Αχμέντ, τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για την Ιεμένη. Επίσης έχουμε πληροφορίες στα μέσα, στα μίδια για συζητήσεις για το ΟΜΑΝ. Ελπίζουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα αποφέρει αποτελέσματα, διότι η Γεμένη έχει έναν πληθυσμό που υποφέρει πολύ, είναι μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση και εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε για να περιορίσουμε αυτή τη σύγκρουση. Θα πρέπει η ύπατη εκπρόσωπος να οργανώσει αυτήν την ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκόμες, το για ένα λεπτό. Βρίσκεται πολύ κοντά στον θρησκευτικό πόλεμο η Εμένη και η διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εντείνουν τι διπλωματικέ προσπάθειε ώστε να υπάρξει η πάυση των εχθροπραξιών το αντίτιμο αν δεν, κάνουμε, αν δεν δράσουμε θα είναι το χάος και κυρίως η καταστροφή της κληρονομιάς της ανθρωπότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι δυνατόν σε σχέση με την ε, κατάσταση αυτή να έχουμε την προώθηση του Ισλαμικού κράτους και θα πρέπει εδώ πραγματικά να υπάρξει αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και να πάψει ο βομβαρδισμός και τα πάνδυνα των αμάχων και που πάσχουν ε, ε, από την πείνα και την ε, ασυτεία. Πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ε, τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες οι διπλωματικές των Ηνωμένων Εθνών για μια προσπάθεια ειρήνης. Ταυτόχρονα η ύπατη εκπρόσωπος Μογκερίνη θα πρέπει να απαιτήσει από τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους κανόνες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγωγή όπλων και εξοπλισμών προς αυτή την περιοχή που, ασκούνται, που ασκεί βία αυτό το φαινόμενο κατά των αμάχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye με τέσσερι παρεμβέσει. Πόλτσακ Καταρχά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αποτίσω φοροτιμής και να εκτιμήσω το γεγονός ότι τα γειτονικά κράτη έχουν υποδεχθεί πρόσφυγες και προσπαθούν να βοηθήσουν. Είναι σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό, διότι κάποιες, κάποιοι ισχυρισμοί μπορούν έτσι να αντιμετωπιστούν, που ακούγονται πολλές φορές όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση στην ίδια τη χώρα, την Ιεμένη, Πρέπει φυσικά η ανθρωπιστική αυτή κρίση με τα πιο κατάλληλα μέσα, διπλωματικά μέτρα και μέσα να αντιμετωπιστεί. Αλλά και ανθρωπιστικά πρέπει να δράσουμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίε, οι σειράξει και από πλευρά των επαναστατών, των εξεγερμένων και των δυνάμεων τη Αλκάιντα, αλλά επίση και των στρατιωτικών δυνάμεων τη Συμμαχία υπό την Σαουδική Αραβία. Πρέπει με διπλωματικά μέσα και μέτρα να προσπαθήσουμε την κυβέρνηση στην Ιεμένη να την καλέσουμε να διεξαγάγει συζητήσεις με όλες τις ομάδες. Ευχαριστώ. Φρουντζούλικα τώρα για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Εμένη βρίσκεται στο χείλος της πιο σημαντικής κρίσης αυτή τη στιγμή εξαιτίας του ότι δεν έχει πρόσβαση κυρίως σε ενέργεια και άλλους πόρους δεν έχουμε να κάνουμε τόσο πολύ με μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο βασικές πλευρές του Ισλαμισμού. Πάντως, ελοχεύει ο κίνδυνος της γενικότερης αποσταθεροποίησης στις περιοχές και βλέπουμε ότι η πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση, η κατάσταση ασφάλειας επιδεινώνονται στην Ιεμένη και αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη περιφερειακή ένταση και ακόμα σε έναν ευρύτερο πόλεμο στην όλη περιοχή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία βλέπουμε ότι θα πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα με την κατάσταση στην Ιεμένη. Δεν μπορούν να χάνονται όλο και περισσότερες ζωέ. Συμφωνώ λοιπόν με τη στάση των ΗΠΑ για να σώσουμε όσο δυνατόν περισσότερε ζωέ και για την εμπλοκή όλων των πλευρών στη δικασία εξέβρεση μια λύση. Θα πρέπει και εμεί να εμπλακούμε και να συνεργαστούμε με όλε τι πλευρέ προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κρίση. Συμφωνώ λοιπόν με τι προσπάθειε των ΗΕ και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμένη ανθρωπιστική δράση προκειμένου να βοηθήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη στην προσπάθειά του για την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια. Νομίζω επίσης ότι οι διαπραγματεύσει μπορούν να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη λύση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε κυριαρχία και εδαφική ενότητα για το σύνολο τη Ιεμένης. Ο κύριο Μαριάς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η κατάσταση στην Ιεμένη παραμένει έκρηθμη και επικίνδυνη, με τη χώρα να βυθίζεται στο χάο. Κύριε Επίτροπε, παρακολουθώντας και διαβάζοντας τον τύπο το τελευταίο εξάμεινο, ο απολογισμό στην Ιεμένη είναι ο εξής Ένοπλε συγκρούσει, αιματοχυσία, στρατιωτική επέμβαση εκ μέρους της σαουδικής αραβίας ναυτικός αποκλεισμός απομάκρυνση του προσωπικού του οηε και των ξένων διπλωματών για λόγους ασφαλείας διώξεις λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων. μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση πείνα ασυτεία χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν για να γλιτώσουν και πηγαίνουν στις γειτονικές περιοχές ταυτόχρονα συγκεντρώνονται γιατί θέλουν να φτάσουν στην ευρώπη ακόμη και στην ελλάδα πλέον έχουμε πρόσφυγες από την ιεμένη. ταυτόχρονα επωφελούνται από αυτή την κατάσταση οι τζιχαντιστές. επομένως το ερώτημα κύριε επίτροπε είναι τι κάνει η ευρωπαϊκή ένωση. όπως ανέφερα και χθες σε άλλη ομιλία μου η στενότερη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως ο οασε και ο ΙΕ θα μπορούσαν να βοηθήσουν να επέλθει η ομαλότητα στην ιεμένη. χρειάζεται πολιτική λύση για την ιεμένη. ευχαριστώ τώρα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά ίσως πρέπει να δώσετε το λόγο στην κυρία Μπιλμπάο, γιατί έχετε δώσει μόνο ένα λεπτό στους φιλελεύθερους. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορείτε να δώσετε το λόγο στην κυρία Μπιλμπάου, η οποία ζήτησε το λόγο και πριν από μένα. Ε, Μα δεν, δεν, δεν ζήτησε το λόγο κυρία Μπιλμπάου, εγώ δεν το βλέπω μπρο στα χαρτιά μου λέει ο πρόεδρο. Πάντως και σε εσά μπορώ να δώσω το λόγο, ενδεχομένω μετά από την κυρία Μπιλμπάου λέει ο μιλητής. Όχι, όχι, πάρτε εσεί τώρα το λόγο, εσεί καλύτερα. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι αντιμετωπίζουμε μία ακόμα απίστευτη ανθρωπιστική κρίση. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Η κατάσταση που έχουμε σήμερα στην Ιεμένη δεν πρόκειται μία νυχτή να διευθετηθεί. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ στρατιωτικέ επεμβάσεις, έχουμε πολλέ παραστρεωτικέ οργανώσει και ομάδε που δραστηριοποιούνται στην Ιεμένη. Μιλάμε για απόλυτο χάο. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μία ακόμα πρόκληση. πώ θα καταφέρει να δώσει την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτή τη χώρα. Διαφορετικά εκατομμύρια ανθρώπων, εκατομμύρια παιδιών θα λιμοκτονήσουν. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα αναγκαστούν να εκτοπιστούν ή θα χάσουν τη ζωή τους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές να έρθουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αυτό από μόνο του μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ότι σιγά σιγά θα αποκλιμακωθεί ο πόλεμος και κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε μια τόσο μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Λοιπόν, έχετε κι εσεί ε, το λόγο για ένα λεπτό, εφόσον είμαστε στη διαδικασία κάτι διάρκεια ούτω ή άλλω. <clears throat> Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αλλά στην αρχή το είχα ζητήσει και λυπούμε αν υπήρξε κάποια, κάποιο λύστημα. Η εμένη εδώ βλέπουμε ότι ένα από τα πιο φτωχά κράτη του κόσμου εμορραγεί ε, ε, και βλέπουμε ότι έχει φτάσει σε αφόρητα επίπεδα ε, η κατάσταση εκεί. Μικρά παιδιά που είναι στρατιώτες, ανθρωποεμπόριο, επιθέσεις σε σχολεία και σε νοσοκομεία και γι' αυτό υποστηρίζουμε άμεσα μια πάυση των εχθροπραξιών, ανθρωπιστική εκεχηρία δηλαδή, για να μπορέσουμε να παράσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Και επιτέλους αυτή η σύραξη να σταματήσει που κρατάει εδώ και δεκαετίες και να υπάρξει μια ε, διεθνής ανάκριση και διακρύβωση τι έγινε με τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Πρέπει ενεργά να δραστηριοποιηθούμε για την ανασυγκρότηση της, χα... χώρας και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε του κατοίκους με κάθε τρόπο και για τους τουρίστες Βάσκους και Καταλανούς ε, που σκοτώθηκαν πριν από χρόνια σε μια επίθεση στη χώρα αυτή θα πρέπει πραγματικά να δούμε πόσα χρόνια διατηρείται αυτή η σύραξη και τι έχει προκαλέσει. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε συζήτηση. Ο κύριος, ο Επίτροπος Χάν έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ευρωβουλευτές, όπως είπα προηγούμενα, όλοι συμμεριζόμαστε τους ίδιους στόχους. Την πάυση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και το να ξεκινήσουν μέσω των Ηνωμένων Εθνών οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων σε χρονική συγκυρία όλο και μεγαλύτερων εχθροπραξιών αυτή η χώρα θα πρέπει να μην διολυστήσει στο χάος και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Βοηθώντας να υπάρξει και χειρία θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής βλέπουμε ότι οι Ιεμενίτες ε, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των κατοίκων της ε, κοινωνίας της Ιεμένης θα μπορούν να προσφέρουν μια αηφόρο λύση σε αυτή την κρίση. Είμαι πεισμένος ότι τα βήματα αυτά θα πρέπει να συμφωνηθούν άμεσα. Άμεσα με μια εκεχηρία για ανθρωπιστικούς στόχους, άμεσα εκεχηρία, ώστε να μπορέσουν να εμπλακούν όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σημαντικό οι διεθνείς οργανώσεις να μπορέσουν να παράσχουν το, την επισητιστική βοήθεια και τα, το ιατρικό υλικό, ιατροφαρμακευτικό υλικό στους κατοίκους της Ιεμένης και να μπορέσουμε να δράσουμε διότι αν δεν υπάρξουν αυτά τα βήματα για την αποκλιμάκωση η σύραξη αυτή έχει πολύ μεγάλο αρνητικό δυναμικό με τεράστιες αρνητικές δυνατότητες για όλη την περιοχή για το κέρα της Αφρικής και στέλος εις βάρος της Ευρώπης. Ήρθε η χρονική στιγμή όλοι να ξαναξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία διαπραγματεύσεων χωρίς όρους και προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει η νόμιμη πολιτική αρχή της χώρας να λειτουργήσει υπέρ των πολιτών. Είναι κοινή ευθύνη όλων των ε, κομμάτων και των εμπλεκομένων στην Ιεμένη και υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας να εργαστούν προς αυτό το στόχο. Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> στεναρά δεσμεύεται ώστε να συνεισφέρει υπέρ αυτής της διαδικασίας όπως περνάει από το χέρι της. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, αλλά θα μείνετε μαζί μας και για την επόμενη συζήτηση. Έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφίσματος ε, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση αυτή, η οποία κλείνει και περνάμε